Ευχαριστώ. Ο George Orwell και ο ίδιος θα έμενε έκπληκτος ε, από το όνομα αυτό. Και μάλιστα δίνουμε σε μια εξαιτία 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ Πολύ ενδιαφέρον. Το ταμείο αυτό που μπορεί να δίνει όπλα σε αφρικανικές χώρες με ιστορία πολιτικών ταραχών, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα τους υποστηρίζει και με στρατιωτική και τεχνική βοήθεια. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος και αν προχωρήσει αυτό το εγχείρημα να αλλάξει όνομα και να ε, ονομαστεί Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για τη Διευκόλυνση των ε, Όπλων ε, Μαλή και Σομαλία. Τα ξέρει κυρία Μογγερίνη. Κοιτάξτε τι έγινε στο Μαλή από τις ε, διάφορες ένοπλες ομάδες που στηρίζουν κυβέρνηση. Εμείς οι Ιρλανδοί ήρθαμε εδώ για να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαφυλάξουμε την ουδετερότητά μας. Δεν διαφυλάσσουμε την ουδετερότητά μας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υποτίθεται ειρηνικό εγχείρημα. Τώρα δεν είναι πια έτσι, δεν είναι. Ευχαριστώ κύριε Φλάναγκαν για να τελειώσει η διαδικασία του Κατσέα. Ο κύριος Παπαδάκης, παρακαλώ. Με τις ευλογίες του Ευρωκοινοβουλίου τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Ο Μπρέχτ από πολύ παλιά σας απαντά όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος γιατί αυτός ο νέος αντιδραστικός μηχανισμός έχει ως αποστολή του την απευθείας χρηματοδότηση χωρίς καθυστερήσεις των στρατιωτικών σωμάτων για υπερελιστικές επεμβάσεις της ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεών της όπου γιατί διπλασιάζει τις στρατιωτικές δαπάνες για τέτοιες αποστολές φτάνοντάς τες στο ένα πέντε δις ετησίως γιατί προκλητικά μάλιστα στο όνομα της ισότητας κάνει προσκλητήριο πολέμου ειδικά στις γυναίκες προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτές τις επικίνδυνες για τους λαούς αποστολές. 70 χρόνια από την ίδρυση του νατο 20 χρόνια από την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ευρωπαϊκής ένωσης 20 χρόνια από τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς γιουγκοσλαβίας από το νατο στείνεται μηχανισμός συστηματοποίησης των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. οι λαοί με την από κοινού πάλη τους να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο τα μονοπόλια το σύστημά τους τι υπερελιστικές ενώσεις και τις κυβερνήσεις τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδάκη. Τελειώνει η διαδικασία Κατσιάη για να κλείσει και η συζήτηση. Ε, εσείς πάλι κύριε Επίτροπε, εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Κίνγκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους βουλευτές που πήραν το λόγο για τις παρεμβάσεις τους, για τις προτάσεις τους. Να πω προς τον κύριο Πιμέντα Λόπες ότι δεν κρύβουμε τίποτα. Ίσα ίσα, είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται. Η έκθεση το αναγνωρίζει. Είναι σαφές τι μέσα θέλουμε, ποια θα είναι η διαδικασία λήψη αποφάσεων και όλα αυτά θα είναι αντικείμενο λογοδοσίας από όποιον είναι αρμόδιος. Η σχετική δουλειά έχει ξεκινήσει σε αρκετούς από τους τομείς, όπως και η έκθεση σωστά αναφέρει. Όπως για να βεβαιωθούμε ότι μελλοντικέ μεταφορές ευαίσθητου εξοπλισμού θα γίνεται με, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και ό,τι άλλο χρειάζεται. Βεβαίω αυτό θα δώσουμε πρώτη προτεραιότητα και επίση συμφωνώ απολύτω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο, πλήρω ενήμερο και συστηματικά για τη χρήση αυτών των, εξοπλισμών. αυτό ακριβώς ε, θα επιζητούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ λοιπόν όλους ε, και ελπίζω η έκθεση να εγκριθεί αύριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Κίνγκ. Για να κλείσει η συζήτηση και πάλι για ένα λεπτό, η κυρία Βότμανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ συχνά άκουσα τη λέξη ειρήνη, ειρήνη και ασφάλεια. Δυστυχώς όμως αυτές οι έννοιες είναι άγνωστες για πολλοί κόσμο στη γη μας. Ξέρουμε παντού ότι έχουμε εμπόλεμες σειράξεις. Γι' αυτό ε, έχει σημασία να έχουμε ένα ευέλικτο μηχανισμό και να μπορούμε ε, να δρούμε πιο αποτελεσματικά διεθνώς, ε, να υποστηρίζουμε τους εταίρους μας και τους συμμάχους μας για να επιμερίζουμε το κόστος. Άκουσα πολλά επιχειρημάτα που δεν έχουν καμιά σχέση με το θέμα μας αυτό το μέσο, το μηχανισμό το χρειάζεται η Ευρώπη για να είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό μας ζητούν και οι πολίτες. Για να μην μας λένε ότι στην εξωτερική πολιτική γαυγίζουμε αλλά δεν δαγκώνουμε. Με αυτό το μηχανισμό επιτέλους μπορούμε να αλλάξουμε τις καταστάσεις επιτρόπου και να ε, υποστηρίζουμε την ειρήνη. Και ελπίζω αύριο να υπερψηφιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βότμαν. Τελειώνει η συζήτηση εδώ και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Η επόμενη συνεδρίαση αρχίζει αύριο στις 9 έχει ε, διανεμηθεί, δημοσιευθεί η ημερήσια διάταξη και μπορείτε να τη βρείτε και στην ισοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, καλή σας επιστροφή. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες και σας εύχομαι μια ευλογημένη και ήσυχη νύχτα. Λήξη συνεδρίασης.